Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι πρόσφατες ε, καταδίκες σε θάνατο ε, χριστιανών που βρέθηκαν ένοχοι βλασφημίας κατά του προφήτη Μοχάμετ είναι πραγματικά πίστευτες ε, και απαράδεκτες. Ακόμη και SMS θεωρήθηκαν ε, αρκετά για κατηγορίες. Είχαμε μαζικές ε, διώξεις των χριστιανών που δεν μπορούν να ασκήσουν τις θρησκευτικές δραστηριότητες. Επίσης, πολύ συχνά έχουμε ε, εμπρισμούς σπιτιών χριστιανών, εκκλησιών, είναι, ενώ οι τοπικές αρχές θελοτυφλούν. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό ότι στον κόσμο που ζούμε που έχουμε τέτοια πολυμορφία πολιτιστική και θρησκευτική, έχουμε αντίστοιχα τέτοιες παραβιάσεις ε, δικαιωμάτων. Στο Πακιστάν δυστυχώς, δεν είναι η εξαίρεση. Πολλέ ε, τέτοια περιστατικά έχουμε και σε άλλες Ισλαμικές χώρες. Με βάση την ε, οργάνωση Open Doors, τελευταία χρονιά δυστυχώς, ενισχύθηκαν και οξύνθηκαν η διώξη χριστιανών στο Πακιστάν που πέρασε από τη 14η στην 8η θέση των χωρών που περισσότερες τέτοιες καταπιέσεις ασκούν. Και μάλιστα στο Πεσαβάρ ε, είχαμε τον ε, Ιούνιο 88 θύματα από εμπρισμό εκκλησίας. Ε, θα ήθελα να απευθυνθούμε στις πακιστανικές αρχές να σταματήσουν αυτές τις παραβιάσεις, να αναθεωρήσουν τους νόμους περί και να εξασφαλίσουν ίσα δικαιώματα σε όλους τους πακιστανούς πολίτες γιατί οι δυσανάλογες ποινές ε, δεν συνάδουν με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και πραγματικά τέτοιες αυστηρές ποινές για, ε, για την περίπτωση πλασμιμίας ε, αντιβαίνουν στις, στο, στο δίκαιο. Ευχαριστώ κύριο Σρέπο. Για ένα λεπτό. Arvoisa puhemies, Pakistanissa on ollut voimassa laki Jumalan pilkassa jo lähes 30 vuotta viime kuukausien aikana pakistanissa on annettu lukuisia kuolemantuomioita jumalan pilkkalain nojalla ja useat tapaukset ovat Το θέμα εδώ πέρα είναι πως υπάρχουν διώξεις ε, τοπικές ε, και κυρίως ε, βεβαίως τα αποτελέσματα τα υφίστανται οι θρησκευτικές μειονότητες. Επίσης και ο ΙΕ ζήτησε να αλλάξει αυτός ο νόμος η ελευθερία του λόγου είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και περιορίζεται μόνο αν υπάρχουν εξαιρετικές καταστάσεις, ε, δηλαδή να υπάρχει ξέρω, πρόθεση θρησκευτικού μίσους, αλλά δεν είναι δυνατόν να κρίνει το κράτος πώς θα σκέφτονται οι άνθρωποι και να ακολουθεί τα όσα λένε οι εξτρεμιστές. Ε, δυστυχώς το ζήτημα αυτό των θρησκείων έχει γίνει πλέον παγκόσμιο πρόβλημα. Οι Πακιστανοί πολίτες πρέπει να έχουν την δυνατότητα να διαμορφώσουν γνώμη. Μια κοινωνία η οποία συζητά είναι πιο πλούσια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Κόρολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω εργαστεί στο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βλέπω πως ε, συχνά το θέμα είναι ερμηνεία των νόμων. Ε, το Πακιστάν είναι μαύρη τρύπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν είναι δυνατόν ας πούμε, να υπάρχουν αυτές οι ποινές ε, ή ένα ζευγάρι χριστιανών που κατατάθηκε καταδικάστηκε σε θάνατο για προσβολή ενός ιερού κειμένου, κάτι το οποίο ήδη αρνούνται. Έχω συναντήσει πολλούς τέτοιους ε, ανθρώπους στο Πακιστάν που κινδυνεύουν με εκτέλεση. Δεν έχει ούτε μία σχέση δε με βλασφημία. Ο νόμος χρησιμοποιείται για λόγους επιχειρηματικούς ή άλλους. Μην ξεχνάμε υπήρχε και ένας υπουργός που, υπήρχε ένας υπουργός που ήθελε να καταργήσει τον νόμο αυτόν περί βλασφημίας ο οποίος όμως δολοφονήθηκε όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Σας ευχαριστώ. Σάκε. Yes. <laughs> Thank you, President. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, συνάδελφοι, οι νόμοι κατά τη βλαστημία στο Πακιστάν ε, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που ονομάζουμε εμεί τα μελιώδη δικαιώματα. Οι μειονότητε υποφέρουν από την εφαρμογή αυτών των νόμων με πολύ ψηλέ ποινέ καταδίκε. Οι νόμοι τη βλασφημία δεν επιτρέπουν την ελευθερία έκφραση σε τέτοιο βαθμό που από τη χώρα ζητήθηκε από του μηχανισμού προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ να καταργηθούν αυτοί οι νόμοι. Επιπλέον, εκατοντάδε εγκλήματα τιμή έχουν ε, διαπραχθεί κατά παράβαση του δικαίου, του διεθνού δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα έδωσε το καθεστώ ε, τη ε, χώρα GSP με τα με τις γενικευμένες δεσμολογικές προτιμήσεις στο Πακιστάν, κάτι που δεν θα έπρεπε να συμβεί. Η κυβέρνηση θα έπρεπε το de facto μορατόριο για τη θανατική καταδίκη να το, να το μετατρέψει σε μια πραγματική κατάργηση τη θανατική καταδίκη και να επιτρέψει την ελευθερία έκφραση. Όχι αυτό να απαγορεύεται για λόγου θρησκευτική μυσαλλοδοξία. Επίση να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ε, προκειμένου να εφαρμοστούν όλοι οι νόμοι κατά τη τρομοκρατία σωστά και να μην παρεμποδίζονται με οργανώσει. Σας ευχαριστώ. Σόζα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι είναι δεκάδες ε, οι περιπτώσεις βίας ε, στο Πακιστάν με αστάθεια για ολόκληρη την γεωγραφική ζώνη και το ίδιο το κράτος του Πακιστάν. Υπάρχουν πολλές θρησκευτικέ μειονότητες στο Πακιστάν και μεγάλη καταπίεση. Και είναι πολλές οι χριστιανέ οι οποίε έχουν αντιμετωπίσει καταδίκες Μιλάμε για διακρίσεις ε, που γίνονται σε καταστάσεις ε, ε, με εξοδικαστική κρίση των υποθέσεων και χωρίς δίκαιη εξέταση. Πολλοί δημοσιογράφοι έχουν χάσει τη ζωή τους, το ίδιο και οι συνδικαλιστέ. Σε αυτό το πλαίσιο, οι γυναίκε είναι ακόμα μια πιο ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού. Το θέμα τη θρησκεία πολλέ φορέ έχει χρησιμοποιηθεί για πολιτικέ σκοπιμότητε. Η θανατική καταδίκη συνεχίζει να ισχύει και πολλέ ε, οργανώσει για τα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν υπολογίσει σε 8.000 τα άτομα που έχουν καταδικαστεί για τέτοιου λόγου σε θάνατο. Μιλάμε για ένα κράτο το οποίο δεν προστατεύει σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα των μειονοτήτων και προωθεί τη βία. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του Πακιστάν να λάβει μέτρα που θα επιτρέπουν την ε, ελευθερία εξάσκηση των θρησκευτικών, πιστεύω, ή τουλάχιστον την ελευθερία τη έκφραση και μέσω του διαδικτύου. Είμαστε μεταξύ αυτών που πιστεύουμε στην δύναμη και τη σημασία τη δράση των όσων βρίσκονται στην ίδια τη χώρα, του άνδρε και τι γυναίκε που αυτή τη στιγμή φημώνονται. Και πρέπει να, και πρέπει να του επιτρέπει να αγωνιστούν για την αλλαγή αυτή τη κατάσταση και τα δικαιώματά του. Ευχαριστούμε. Κρόνμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η θρησκευτική βία συνεχίζεται στο Πακιστάν. Καταδικάζουμε δρυμύτατα όλες τις ε, βαναυσότητες κατά θρησκευτικών κοινοτήτων, καθώς και τις διακρίσεις και την μυσαλλοδοξία ε, λόγω θρησκείας ε, ή δοξασίας και ομολογίας. η δοξασιας και ομολογιας κυβέρνηση του Πακιστάν θα πρέπει να προστατεύσει τα θύματα παρενοχλήσεων και θρησκευτική βία, να μην ε, ενισχύσει η ρητορική μίσου και να προαγάγει την ανεξιθρησκεία και την αμοιβαία κατανόηση. Θα πρέπει επίση να διωχθούν οι δράστες της ε, ε, επιβολής των καταγγελιών βλασφημία και των εξυμνών των μίσους. Επίσης θα πρέπει να, να τροποποιηθεί ο αντιτρομοκρατικός νόμος και η σχετική νομοθεσία για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ακολουθούν οι ομιλητέ ξενόμενων των ομάδων. Πόσελτ, για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, το Πακιστάν έχει δύσκολη ιστορία. Πρόκειται ακόμα και το όνομά του. δε είναι τεχνητό, όπως και η χώρα είναι τεχνητή, καθώς οι Βρετανικές Ινδίες ε, μοιράστηκαν σε ε, μια Ινδουιστική χώρα με μουσουλμανική μειονότητα και μια μουσουλμανική χώρα με Ινδουιστική μειονότητα. Και αυτό μέχρι σήμερα έχει φοβερές συνέπειες, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε απλούστατα να, υπάρξει, ε, να υπάρχει αυτή η βία όχι μεταξύ μόνο Ινδουιστών και Μουσουλμάνων, των διαφόρων ομολογιών του Ισλάμ, αλλά ειδικά κατά των χριστιανών. Και αγαπητοί συνάδελφοι, θα το πω ξεκάθαρα, οπωσδήποτε είμαστε υπέρ της όλων, αλλά ποιος θα ζητήσει την προστασία των χριστιανών, εάν όχι εμείς οι Ευρωπαίοι. Είναι βασική μας αποστολή, την οποία πρέπει να στην οποία πρέπει να ανταποκριθούμε και ε, έναντι του Πακιστάν. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Μέσερσμιτ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, πρέπει να έχουμε υπόψη ότι αυτά που συμβαίνουν στο Πακιστάν είναι σημαντικά. Πρέπει να δούμε τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σε αυτή την ε, προσπάθεια πρέπει να σκέψουν όλοι οι συνάδελφοι. Δεν είναι καινούργιο το θέμα φυσικά. Έχουμε ξανασυζητήσει τέτοια, επίπεδα, τέτοια θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, το ε, Συμβουλίο των Υπουργών πιστεύω ότι θα πρέπει να αναλάβει δράση. Εμεί είμαστε απλοί βουλευτέ, πρόσωποι των πολιτών και δεν είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τέτοιε καταστάσει. Είδαμε κάτι ανάλογο να συμβαίνει και στην περίπτωση τη Ουκρανία αλλά και στο Πακιστάν. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για το Πακιστάν είναι να ζητήσουμε από τι εθνικέ μα κυβερνήσει να αναλάβουν ε, εκείνη δράση. Παρά να ζητούμε από έναν κακομίρι επίτροπο που δεν μπορεί να κάνει και πολλά εδώ να αναλάβει δράση εκ μέρου μα. Όχι, θα πρέπει οι εκλεγμένε κυβερνήσει να αναλάβουν τι ευθύνε του και ε, όχι εμεί εδώ να συζητάμε για τέτοια θέματα. Στο ημικύκλιο που είναι ούτω ή άλλω και άδειο. Ευχαριστώ. Κέλλη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ με τους συναδέλφους μου όταν μιλάμε για την καταδίκη των νόμων περί του Πακιστάν και πράγματι αυτή ήταν η κατάσταση ακόμα και πριν ιδρυθεί το Πακιστάν το 1947 αλλά το 1980 ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο οι νόμοι αυτοί και εισήχθη η θανατική ποινή για τη βλασφημία. Μετά το 2013 καταδικάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για βλασφημία και υπάρχουν αυτή τη στιγμή 17 άτομα που αναμένουν εκτέλεση και άλλοι 20 ε, που έχουν καταδικαστεί σε ισόβια. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να τερματιστεί αυτή η κατάσταση, ειδικά όσον αφορά την εισαγωγή ενός νέου τρόπου σκέψης στο Πακιστάν. Ε, Κύριε Κέλλη, δέχεστε ερώτηση από τον κύριο Πόσελτ. Ε, Κύριε Πόσελτ, στον κύριο Σμιτ εγώ ήθελα να απευθύνω ερώτηση. Όλος εξαιρετικός. Κύριε Σμιτ συμφωνείτε? Ναι, ναι, ναι, είπε ναι. Ωραία. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο Σμιτ γιατί χρησιμοποιεί αυτό το σημαντικό θέμα για να επιτεθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μη Κομισιόν νομίζω κάνει εξίσου καλή δουλειά όπως και οι εθνικές κυβερνήσεις. Απλά έχει περισσότερο βάρος γιατί εκπροσωπεί ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο ένα κράτος. Øh, er- Όταν συγκρίνουμε αυτά που έχει κάνει η Λέδια στον εδώ και πέντε χρόνια με αυτά που κάνουν οι κυβερνήσεις, αλλά να με συγχωρείτε, δεν υπάρχει καμία σχέση. Είναι σαφές ότι σε όλες τις ε, περιπτώσεις όταν βλέπουμε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν οι κυβερνήσεις να πετυχάνουν αποτελέσματα όπως συνέβαινε ανέκαθεν εδώ και αιώνες άλλωστε. Ε, εδώ από τότε που ιδρύσαμε αυτή την ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ουσιαστικά διασπαθίζουμε δημόσιο χρήμα και δεν υπάρχει και καμία νομιμότητα στη δράση αυτής της υπηρεσίας. Περνάμε στο Catch έχουν ζητήσει πάρα πολύ το λόγο. Γι' αυτό θα λάβουν υπόψη και άλλα καρτήρα προ το ποιος μιλάει πιο συχνά. Λοιπόν, η κυρία Γέγκλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Τα γεγονότα και οι αποφάσεις των δικαστηρίων στο Πακιστάν για βλασιμία είναι απίστευτα αυστηρές. Η προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων είναι βασική κατευθυντήρια γραμμή της εξωτερικής μας πολιτικής. Οι χριστιανοί είναι πάντα στόχοι διακρίσεων παγκοσμίω. Εδώ πέρα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά. Οποιαδήποτε μορφή εξτρεμισμού είναι καταδικαστέα. Ειδικά σε μια σημαντική χώρα όπως το Πακιστάν, το οποίο θεωρεί αυτόν ε, περιφερειακή δύναμη. Ε, πρέπει να αποτελεί υπόδειγμα κράτους δικαίου, ειδικά δεδομένης της κατάστασης στο Αφγανιστάν. Μόνο εάν καταπολεμήσουμε από κοινού τις ε, ακρότητες θα μπορέσει να σταθεροποιηθεί το Πακιστάν και έτσι θα ωφεληθεί όλη η περιοχή όλη η κεντρική Ασία θα μπορούσε να αποτελέσει ένα λαμπρό παράδειγμα και αυτός πρέπει να είναι ο πολιτικός μας στόχος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μετά από 15 χρόνια αυτή ήταν η τελευταία μου ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία. Καλή δύναμη ε, ευχόμαι στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ και σε εσά ε, καλή συνέχεια. Κυρία Γκουρμάη. Ευχαριστώ. Οι πρόσφατες διώξει εξαιτία βλασφημίας η συμμετοχή σε θρησκευτική μειονότητα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικέ. Και παρά τα μέτρα που έλαβε η πακιστανική κυβέρνηση το 2008, η καθημερινή κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων είναι ιδιαίτερα επισφαλής και όπω φαίνεται από το ψήφισμα έχουμε σοβαρότητες και κατάφορες παραβιάσεις ελευθερία, συνείδηση, ε, σκέψη και θρησκείας. Επίση, έχουμε αναγκαστικούς γάμου κοριτσιών και γυναικών. Αυτό είναι απαράδεκτο και οι σχετικέ δολοφονίε. Η πακιστανική κυβέρνηση θα πρέπει σοβαρά να αυξήσει τι προσπάθειε τη ε, και να αντιμετωπίσει, να Καταρχήν να τροποποιήσει την νομοθεσία ε, και να προληφθούν τα εγκλήματα κατά θρησκευτικών μειονοτήτων, αλλά και οι διώξεις, ε, να γίνουν διώξεις των δραστών αυτών των εγκλημάτων. Επίσης, ό,τι αφορά την κατάσταση των γυναικών, θα πρέπει να βελτιωθεί η κατάστασή τους ε, και η πρόσβασή τους στην παιδεία, ξεκινώντας από τα θρησκευτικά σχολεία, τους μετρεσέδε. Αλλιώς, ολόκληρες γενιές κοριτσιών και γυναικών θα πάνε χαμένες. Σα ευχαριστώ. Κυρία Χίμπνερ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, έχουμε να κάνουμε με μια χώρα που ε, εφαρμόζει ένα ανήκουστο δίκαιο, το δίκαιο του θανάτου, ε, για λόγους βλασφημίας κατά του προφήτη Μωάμεθ. Πουθενά σε κανένα άλλο κράτος του κόσμου άνθρωποι που λένε κάτι κακό για τον προφήτη ή μπορεί ένας γείτονας να καταγγείλει τον γείτονά του έστω και ψευδός και να το συκοφαντήσει γιατί έτσι πραγματικά παραβιάζονται κατάφορα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει όλοι να πούμε στεναρά όχι, φτάνει πια. Εμείς δεν αναγνωρίζουμε τέτοιο δίκαιο, δεν ανεχόμαστε τέτοιο δίκαιο. Αυτή τη στιγμή ε, η χώρα αυτή επιβάλλει περιορισμού σε όλες τις θρησκευτικέ κοινότητες και μειονότητες. Είναι εκτεθειμένοι ιδιαίτερα οι χριστιανοί που δεν μπορούν να, να, να, ασκήσουν τη θρησκευτική του λατρεία. Τέτοιε πρακτικέ στον 21ο αιώνα είναι ανεπίτρεπτε. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ένα χειρό όχι στο Πακιστάν. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Επίτροπος έχει το λόγο για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν είναι πραγματικά στην πρώτη γραμμή των ε, μεριμνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το έχουμε επισημάνει στην κυβέρνηση του Πακιστάν. Έχουμε τονίσει την ε, ανησυχία μα για το κλίμα ε, μεσαιροδοξία και βία, για τι χριστιανικέ μειονότητε, για του Ινδουιστέ, για του νόμου του οποίου αναφέρατε εσεί κατά τη βλασφημία. Εδώ το θέμα είναι ότι στο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα Ευρωπαϊκή Ένωση Πακιστάν και πολύ πρόσφατα είχαμε την παρέμβαση τη υπέτη ε, εκπροσώπου κυρία Άστον ε, που μίλησε με τον ε, σύμβουλο των θέματων αυτών του Πακιστάν, τον κύριο Αζή. Και ο κύριος Λαμπρινίδη, ο ειδικό αντιπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα παρέμβει και για το θέμα αυτό προκειμένου να επιρρώσει τι θέσει μα και θα πρέπει οι εκτελέσεις του Πακιστάν να πάψουν διότι δημιουργούν πραγματικά βίαιες συγκρούσεις και περιστατικά σε όλες τις περιοχές της χώρας κατά των θρησκευτικών που και σας αναφέρατε. Επίσης οι γυναίκες εργαζόμενες όπως είπε η κυρία Γκουρμάη που φέρουν από διακρίσεις, οι άνθρωποι που εργάζονται στην εκπαίδευση και την υγεία, στα σχολεία και κυρίως υπάρχει και ένα θέμα με τη θέση των κοριτσιών στα σχολεία. Υπάρχει κατάχρηση τον ε, και παραβίαση συστηματική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρέπει να υπάρξει ένα τέτοιο ε, καθεστώς για την εκπαίδευση και να μην είναι αντικείμενα χειραγώγηση από αδίστακτου πολιτικού ή θρησκευτικού ηγέτε ή άνεργοι ε, Για να επιληθούν αυτά τα ζητήματα, λοιπόν, θα πρέπει να καταβληθούν προσπάθειε από τι αρχέ για να καταπολεμήσουν τη βία και την μισοδοξία, την έλλειψη ενοχή και τα, τις βίες ομάδες που είναι, θα πρέπει να γίνουν αυτές οι πρώτες τους προτεραιότητες. Θα πρέπει να είναι και για την Ευρώπη μια προτεραιότητα αυτό, αλλά και για τη σταθερότητα της ευρύτερης γεωγραφικής ζώνης, να στηρίξει τη μεγάλη πλειοψηφία των ε, Πακιστανών που δεν είναι υπέρ της εξτρεμιστικής ε, βίας, ούτε της, ε, του κατακαιρματισμού της χώρας βάσει των θρησκευτικών πεπιθήσεων. Θέλουν τον εκδημοκρατισμό της χώρας τους. Θα πρέπει λοιπόν και με διάλογο, αλλά και με πρακτική βοήθεια να στηρίξουμε το Πακιστάν σε αυτές τις προσπάθειες. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα πρόγραμμα κατά των, ε, της διακριτικής μεταχείρισης βάσει ομο, θρησκευτική ομολογίας στο Πακιστάν. Θα πρέπει όλα αυτά να διαχειριστούν και μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της εκπαίδευσης και των, ε, των δυνάμεων της τάξης. Θα πρέπει η διακριτική μεταχείριση να πάυσει καθώς και οι επιθέσεις βάσει της Ε, των θρησκευτικών πιστεύω. Και θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένοι μηχανισμοί ε, αντιμετώπιση και αναχέτηση τέτοιου είδου επιθέσεων. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει την πρόσβαση των ευάλωτων ομάδων στη δικαιοσύνη, να βοηθήσει στην ε, επιβολή του νόμου και την ε, οικοδόμηση υγιών ε, δικαστικών οργάνων. Η εκπαίδευση και ο εκπαιδευτικό κλάδο είναι ένα θέμα που μα ενδιαφέρει στη βοήθεια που προσφέρουμε στο Πακιστάν ω Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να υπάρχει ανοχή για όλε τι θρησκευτικέ ομολογίε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά τη συμπερίληψη του Πακιστάν στο γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων απαιτεί την, ε, το σεβασμό των διεθνών συμβάσεων προκειμένου να υπάρξει σταθερή πρόοδος για την ε, προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το θέμα της ε, ανεξιθρησκείας της ελευθερίας έκφρασης θα συνεχίσει να αποτελεί προτεραιότητα. Το ίδιο και η ευθύνη του Πακιστάν για την προστασία όλων των πολιτών ανεξαιρέτως, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών και των υπόλοιπων μειονοτήτων, καθώς και τα δικαιώμα, ο σεβασμό των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών. Για να γίνουν αυτά θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι, κύριε Μέσο Σμιτ. Και ε, η Επιτροπή και το Συμβούλιο και το Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες που πιστεύουν στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σόνικ και από τη διαδικασία. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. Γιατί είμαστε καμιά δεκαριά στην αίθουσα και μια και είναι η τελευταία μας σύνοδος πριν τις εκλογές θα μπορούσατε να παρατείνετε λίγο το κατστιάι και να επιτρέψετε σε όλους όσους ζητούν το λόγο να τον λάβουν. Θα ήταν ευάρεστο πραγματικά να κάνετε δεκτό αυτό το αίτημα. Κύριε Σόνικ, το είπα από την αρχή πως δεν γίνεται. Έχουμε άλλες δύο διαδικασίες και HDI. Δεν έλαβα υπόψη τους άλλους συναδέλφους. Λυπούμε ούτε και αυτή την τελευταία μέρα δεν μπορούμε να, να επιτρέψουμε να διαρκέσει η διαδικασία για πάντα. Τελείωσε λοιπόν η συζήτηση. Υπάρχουν έξι ψηφίσματα. Ισοφορία θα λάβει χώρα μετά την συζήτηση. Μετά έχουμε το θέμα της Συρίας, ε, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται κάποιες πάλι ευάλωτες κοινότητες.